αυτή, αυτό το αίτημα και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή, το αίτημα άρσης ασύλια το FTT, το END ζήτησαν διορισμό κάποιων συναδέλφων τα ονόματά τους θα τα βρείτε και αν μέχρι την έξοδο των πρακτικών δεν εκφραστούν αντιρρήσεις θα, θεωρούν, θα θεωρηθούν εγκεκριμένοι και αυτοί οι διορισμοί.